Il Presidente! Cari colleghi Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχή της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία διεκόπη την Τετάρτη 15 ε, ε, Μαρτίου αλλά που έχει διακοπεί στις Βρυξέλλες ε, εδώ και δύο χρόνια λόγω των εργασιών που έγιναν στην οροφή. Ci sono foto e filmati sui lavori svolti βλέπετε ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ οι εργασίες οι οποίες ε, κατέδειξαν τη δυσκολία του εγχειρήματο αφενός αλλά ε, και το καλό αποτέλεσμα και η θετική τελική έκβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος την ε, διοίκηση, ιδιαίτερος δε τη Γενική Διεύθυνση Κτηρίων για αυτόν τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε με το θέμα. Τα πρακτικά της 13ης ε, ε, Μαρτίου ε, του 2014 είναι στη διάθεσή σας, υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι από ό,τι φαίνεται, επομένως τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφη 3 και 4 του κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Εποθέσεων στην συνεδρία